Good afternoon, colleagues. Καλησπέρα συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρο. Ονομάζομαι ως και είμαι προσωρινό, πολύ προσωρινό πρόεδρο σε αυτήν την συγκρότηση σε σώμα τη αντιπροσωπεία για το ΝΑΤΟ. Και καλώς ορίσατε έναρξη της ε, συνεδρίασης. Ο σκοπός συνεδρίασης είναι να συγκροτηθεί σε σώμα πρώτα-πρώτα το Προεδρείο αυτής της υποεπιτροπής, εκλογή Προέδρου, δύο αντιπροέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 213 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Πρώτα-πρώτα εκλεγούμε τον Πρόεδρο και στη συνέχεια τους ε, αντιπροέδρους ε, και αυτό θα γίνει από τον νεοκλεγέντα Πρόεδρο περίπου 30 λεπτά. Έχουμε στο 4 έχουμε σύντομη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την αντιπροσωπεία ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή στην 65η Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο, ε, στο Λονδίνο στις 11 ε, Οκτωβρίου. Μου είπαν ότι θα, συ, θα συμμετάσχουν στην ψηφορία κάποιοι αναπληρωτέ, η Άτσα Γενικευζιέννη, ο Σάντρα ο Γιώργη Μπούζε και ο Ντέιβιντ Μακάλιστερ για το ΕΛΚ και ο... η Μαζαλή Αγγιλάρ και η Άννα Φωτίγκα για το ECR. Έτσι είναι, μάλιστα. Επίση, ε, πολλέ ομάδε μπορούν να λάβουν τον λόγο πριν αρχίσει η ψηφοφορία και επίση έχουμε αυτό το πακέτο καλωσορίσματο και την έκθεση δραστηριοτήτων από την ε, ε, γραμματεία, το έχετε λάβει και υπάρχει και ηλεκτρονικά στο ίντερνετ αυτή η έκθεση. Άρα, συνάδελφοι, ας εκλέξουμε τώρα τον ή την πρόεδρο. Παρακαλώ η γραμματεία να ε, δει αν υπάρχει η απαρτία, η απαραίτητη, ναι. Σας ευχαριστώ και σύμφωνα με το άρθρο 218 απαρτία είναι ποσόστοση του αριθμού μας. Τρεις δηλαδή. Επίσης σας υπενθυμίζω ότι ο ή υποψήφιος θα πρέπει να προταθεί από μια πολιτική ομάδα ή από το ένα εικοστό των ε, μελών. Έχουμε την απαρτία Οπότε μπορείτε να κάνετε τις προτάσεις σας για τους υποψηφίους. Διαπιστώνουμε ότι το ΕΛΚ έχει προτείνει τον κύριο Κρίς Πίτερς. για να γίνει πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ. Σάντρα για το ΕΛΚ. Με μεγάλη μου χαρά, λέει η Σάντρα, θέλω να προτείνω για υποψήφιο ε, για τη θέση του Πρόεδρου, τον Κρίς Πέτερς. Εξαιρετική υποψηφιότητα, συγχαρητήρια. Κύριε Κρίς Πέτερς, συμφωνείτε? Πέτερς. Ναι, είναι μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ. είναι ε, τακτικό μέλος και έχει συμπληρώσει την ε, δήλωση για τα οικονομικά συμφέροντα και για τη δέουσα συμπεριφορά. Υπάρχουν άλλες ψηφιότητες. Όχι. Άρα, ένας μόνο είναι ο υποψήφιος και προτείνω να ψηφίσουμε διαβοής. Συγχαρητήρια κύριε Πέιτερς. Περάστε να καθίσετε. Okay. First of all, I would Ο πρώτος, πρώτα απ' σας ε, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας και για τη θετική ψήφο. Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι πρόεδρος. Και βέβαια συγχαρητήρια στους προκατόχους μου και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με επιτυχία. Αγαπητοί συνάδελφοι, και τώρα πάμε να ψηφίσουμε τους αντιπρόεδρους ενημερωτικά έχω να σας πω ότι μου είπαν ότι οι εξή αναπληρωτές θα λάβουν μέρος στην ψηφοφορία Ράσο Γιουγνεβιτσένια, ελπίζω πρόθερα στο όνομά σας ε, θα είχαμε την εξάσκηση θα τα πάμε καλύτερα Σάντρα Καλνιέτα Γερζιμπούσεκ και Ντέβιντ Μακάλιστα αλλά επίσης και η Μαζάλη Αγγιλέρ όπως και η κυρία Φωτίγκα. Συμφωνείτε, ναι. Αν θέλετε κάτι να πείτε, πολιτικές ομάδες, πρέπει να το κάνετε πριν την ψηφοφορία. Επίσης να δούμε αν έχουμε απαρτία, μπορεί να το κάνει η γραμματεία, μάλιστα λέει ο γραμματέας, έχουμε απαρτία. Και τώρα, πέστε μου τις υποψηφιότητες για τον πρώτο και δεύτερο αντιπρόεδρο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω την να πρώτη την κυρία Μπομφρισκό για πρώτη αντιπρόεδρο της ε, μα. μας. Επί τρία χρόνια ήταν ε, γερουσιαστής και έχει ασχοληθεί με τον προπολογισμό της άμυνας. Ήδη είναι μέλος ε, στις εξωτερικές υποθέσεις και επίσης στην Υποεπιτροπή ε, Άμυνας. Και οπότε έτσι θα έχουμε μια πρώτη αντιπρόεδρο γυναίκα, κάτι το οποίο ε, αποτελεί απόδειξη ότι τηρεί τις υποσχέσεις της, το, τους στο Κοινοβούλιο. Επίσης να λάβουμε υπόψη τον κανόνα Ντόντ που είναι μια δημοκρατική αρχή για το Κοινοβούλιο και έτσι μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας Ντόντ και στην Επιτροπή μας. Μάλιστα, συμφωνείτε για αυτή την ε, ε, υποψηφιότητά σας. Ναι, ναι, ναι, λέει η υποψήφια. Συμφωνώ. Ζήτησε κανείς το λόγο, εσείς. Ο κύριος Αουστροβίτσιος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Και είναι τιμή μου να προτείνω τη συνάδελφο Ναταλή Λουαζό για τη θέση αυτή. είναι πολύ γνωστή από τα καθήκοντά της, από τις ευτυχισμένες δραστηριότητές της, Ναταλή Λουαζό, λοιπόν. Δύο υποψηφίους, λοιπόν, έχουμε. Θέλει κανείς άλλο το λόγο? Εάν όχι, θα πρέπει να οργανώσουμε τώρα την ψηφοφορία. Μία ψήφος για κάθε βουλευτή και η κατανομή μεταξύ των πολιτικών ομάδων είναι ΕΛΚ 3 ψήφοι, Σοσιαλδημοκράτε 2, Renew 2, Πράσινη 1 ψήφο, ID 1, ECR 1 ψήφο. Προτείνω να ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Α, ζητώ συγγνώμη. Τρέχω. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Λουαζό. Πρέπει να σας ρωτήσω εάν συμφωνείτε με την υποψηφιότητα... Ναι, ευχαριστώ τον Πέτρα Σαουστρεβίσιους, λέει η κυρία Λουαζό, και συμφωνώ με την υποψηφιότητά μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, προτείνω να ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία μόλις είστε έτοιμοι. Okay. Uh, uh, to be very uh, clear and very short. Λοιπόν, για να πάει καλά η ψηφοφορία, μας προτείνει η Γραμματεία τις εξής οδηγίες. Το πράσινο για, πρώτο, για την πρώτη υποψήφια, το, το κόκκινο για τη δεύτερη υποψήφια. Με τις ε, κάρτες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία βεβαίως που είναι απαραίτητες. Κάντε επαλήθευση. Έχετε όλη κάρτα. Oh, wait. Okay. We can, we can start the voting. Okay. We... Αρχίζει η ψηφοφορία. You can see also on the screen. Επτά για τη δεύτερη υποψήφια, ένας για την πρώτη υποψήφια. Συγχαρητήρια. Οι εκλογές είναι εκλογές. Και όταν έχουμε δύο υποψηφίους πρέπει να επιλέξουμε έναν υποψήφιο, άρα συγχαρητήρια κύριε Λουεζό. Then Λοιπόν, τώρα για τη θέση του δευτέρου αντιπροέδρου. Excuse me for the second vice chair. Λοιπόν, για τη θέση του δευτέρου αντιπροέδρου, ένας υποψήφιος ξέρω ότι υπάρχει, μία υποψηφιότητα. Μισό λεπτό να δώσω το λόγο σε εσά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. καταπατείται ο κανόνας Don't σε αυτή την επιτροπή, όπως και σε όλες τις επιτροπές. Ο κανόνας Don't θέλει να δώσει δημοκρατική έκφραση σε όλους τους συμμετέχοντες. Για τη θέση του Δευτέρου Αντιπροέδρου και πάλι υποψηφιότητα της κυρίας Μπονφρίσκο. Παρακαλώ. άλλε υποψηφιότητε. Ως μέλος της αντιπροσωπείας των σοσιαλδημοκρατών σε αυτή την ε, αντιπροσωπεία προτείνω τον συνάδελφο κύριο Μίξερ από την ομάδα των σοσιαλδημοκρατών. Πρέπει να ρωτήσω και τους ιδίους αν συμφωνούν με την υποψηφιότητα. Βεβαίως. Και εσείς για δεύτερη φορά. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία και πάλι. με την ίδια μέθοδο όπως και πριν. Το πράσινο για την κυρία Μπονφρίσκο και το κόκκινο για τον κύριο Μίξερ. Άρχεται η ψηφοφορία. We open the, the vote. Ding. Λοιπόν, λειτουργεί το σύστημα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. The result is uh, that Mr. Um, εκλέγεται ο κύριος Μίξε. Συγχαρητήρια κύριε Μίξε. Θα πω για δεύτερη φορά ότι έτσι λειτουργούν οι εκλογές. Κάποιος εκλέγεται, κάποιος δεν εκλέγεται. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε. Okay. Um, once again, thank you very much. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Πάμε στο σημείο 4, ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Ήδη είπαμε ότι γίνεται η ετήσια σύνοδος του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο, 11 με 14 Οκτωβρίου. Ξέρετε νομίζω τις πιο σημαντικές πληροφορίες για αυτή την ετήσια σύνοδο. Οπότε δεν χρειάζεται να εξηγήσω εγώ τώρα τα πάντα. Βεβαίως αν υπάρχουν ερωτήσεις να απαντήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση στο Λονδίνο. Και επίσης, άλλο ένα σημαντικό σημείο είναι ότι η έκθεση θα δοθεί στις 11 ή 12 Νοεμβρίου για τα αποτελέσματα, τα απορίσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο. Αν έχετε σχόλια, τώρα είναι η ώρα. Να σας ακούσουμε. Όλα ξεκάθαρα. Έχετε ερώτημα, παρακαλώ. Ίσως εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Ζητήσατε ποια είναι τα μέλη της ε, αντιπροσωπείας που θα πάνε στο Λονδίνο. Όχι. Εγώ ξέρω ότι έχει αποφασιστεί η συμμετοχή στην αντιπροσωπεία. Τα μέλη το γνωρίζουν ότι θα πάνε, δηλαδή. Ωραία. Άλλα ερωτήματα ή προτάσεις? Ωραία. Άρα μπορούμε να κλείσουμε τη συνάντηση αυτή. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε σύντομα.